Τα χθεσινά πρακτικά έχουν διανεμηθεί. Έχετε σχόλια για τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Στη συνέχεια έχουμε την ψηφοφορία για την αίτηση διαβούλευσης της Επιτροπής των Περιφερειών σε σχέση με το σχέδιο